Επεξηγήσεις ψήφου λοιπόν επί των ε, συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Άννα. Παρακαλώ να φύγετε από την αίθουσα με ταχύτητα. Και παρακαλώ να επεξηγήσει την ψήφο του. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Πολύ συχνά έχω την αίσθηση ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ωστόσο, η αντίδρασή τους στις πρόσφατες υποβαθμίσεις αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η αντίδραση αυτή είναι αντίδραση νευρωτικού οργανισμού, θεμελιωδός νευρωτικού οργανισμού. Θα έλεγε κανείς ότι θα προσπαθούσαμε να κάνουμε ότι ε, δεν συμβαίνει τίποτα και έτσι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μα δεν μπορούμε να τυποκρινόμαστε. Ο κύριος Έλμαρ Μπρόκ είπε ότι είναι μια αγγλοσαξονική πλεκτάνη για να υποβαθμιστεί η Ευρώπη δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, δεν υπάρχει αναλλακτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν μπορεί κανείς να βελτιώσει το καιρό ε, ε, εκδίδοντας ένα μετρολογικό ε, δελτίο το οποίο να έχει πιο ήπιους τόνους. Εάν σπάσουμε το τζάμι θα μπει η βροχή μέσα ούτως ή άλλως και θα πλημμυρίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριος Φόξ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως προς τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον περασμένο μήνα, θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεγελούμε τους εαυτούς μας εάν νομίζουμε ότι είμαστε η μόνη φωνή δημοκρατίας στην Ευρώπη. Πολλής λόγος γίνεται για την κοινοτική μέθοδο. Ωστόσο, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η διακυβερνητική συνθήκη υπογράφεται από 26 δημοκρατικώς εκλεγμένες κυβερνήσεις οι οποίες είναι υπόλογες στους λαούς τους. Η δική μου κυβέρνηση επέλεξε να μην συμμετάσχει. Νομίζουμε ότι δεν είναι καλό ούτε για την Βρετανία ούτε για την Ευρωζώνη. Τη Της ευχόμαστε όμω κάθε επιτυχία στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων της. Θα έλεγα ότι η συμπερίληψη στο ψήφισμα μίας αναφοράς στο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, ήταν εντελώς εκτό τόπου και χρόνου. Θα έπρεπε να γίνεται λόγος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη και όχι την υιοθέτηση περισσότερων φόρων οι οποίοι ε, λειτουργούν ε, αρνητικά και έχουν δυσμενείς συνέπειες. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος, ε, η συνάδελφος Κολάνης Κραμποβίνσκα έχει το λόγο. Ή βρίσκεται στην αίθουσα? Δεν βρίσκεται. Σπινμπούκ. Βρίσκεται στην αίθουσα, παρακαλώ. Με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούμε, παρακαλώ. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να πω το εξής. Ε, στο πλαίσιο των επεξηγήσεων ψήφου. Για χρόνια ολόκληρα γινόταν λόγος για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επίσης ε, διεξήχθησαν δημοψηφίσματα για την υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας και αντί τώρα να εφαρμόζουμε τις διατάξεις της, βλέπουμε κυβερνήσεις τη Γαλλία και τη Γερμανία μεταξύ άλλων και κυρίως να ε, υπονομεύουν αυτή τη συνθήκη της Λισαβόνας. Στην περίοδο κρίσης που διανύμουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά οπισθοχωρεί κάτι το οποίο είναι πολύ αρνητικό και πολύ επικίνδυνο. Αντί να ενισχύουμε τις κοινοτικέ πολιτικές, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, αντί να δουλεύουμε όλοι μαζί, αυτή τη στιγμή αποσυναρμολογούμε σιγά σιγά ε, το σύστημα και πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή τη τάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ καταψήφισα το ψήφισμα όσον αφορά τη διακυβερνητική. Δεν είμαι κατά του περιεχομένου του, αλλά είμαι κατά του να λάβει μια θέση αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται για μια συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί έτσι από αυτό το σώμα. Η κρίση στην Ευρωζώνη είναι συνεχή και φαίνεται ότι περισσότερε από τι λύσει που προωθούνται ή που έχουν προωθηθεί μέχρι στιγμή μέσω πολύπλοκων κανονισμών και ακόμα πιο σύνθετων ε, χρηματοπιστωτικών δομών δεν έχουν αποτέλεσμα στις ε, αγορές. Νομίζω ότι μια δικαιωματική συμφωνία θα ήταν πιο αποτελεσματική. Ε, αλλά δεν βλέπω καμία αξία σε κάτι, τέτοια, σε κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο σπαταλάει το καιρό του γιατί χάνουμε το χρόνο νομοθετούμε σε αυτό το σώμα. Εάν οι χώρες μέλη δεν μπορούν να εμπιστευτούν η μια την άλλη ε, για να εκπονήσουν μια σαν νομοθεσία, πώς είναι δυνατόν να έχουμε αποτέλεσμα, πώς είναι δυνατόν να μας εμπιστευτούν άλλοι. Ε, η κυρία Γιάτεν Μάκη έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Φοβόμαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά ε, διατυπώνει κάποιους κανονισμούς και κάποιους διαγωνισμούς που τελικά κανονισμούς που δεν τηρούνται. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες, οι κανονισμοί και να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στόχοι είναι τέτοιοι που δεν πιστεύω ότι πράγματι μπορούν να επιτευχθούν από τις χώρες μέλη. Και στη φάση αυτή νομίζω ότι θα ήταν πιο σημαντικό να έχει εγκριθεί ένα πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να εκπληρωθεί. Και πέραν τούτου θα έπρεπε να μπορούμε να συγκεντρωθούμε στην ανάπτυξη και στην διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έλαβε υπόψη τη ότι συνεχίζουν να υπάρχουν φορολογική παράδοση και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Πιατικάνεν έχει το λόγο. Ναι, θεωρώ την ε, θέση του Κοινοβουλίου ως ιδιαίτερα σημαντική γιατί ε, συμπεριλάβει την αξία των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η τήρηση των κανόνων και η τήρηση, η εκπλήρωση της κοινοτική μεθόδου ως τμήμα της δημοκρατικής διαδικασίας. Αν τώρα για πολιτικούς λόγους υποχρεώθηκε κανείς ε, ήταν ε, μάλλον αναγκαστικό να μην μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι χώρες ε, μέλη, το στο χειρότερο. Αλλά σημαντικό είναι να πληρούνται η κοινοτική μέθοδος, όπως έγινε με τη, με τη δέσμη των έξι νομοθετικών μέτρων. Σημαντικό είναι τώρα να τηρηθεί η συνήθις νομοθετική διαδικασία κατά την εφαρμογή αυτών των νέων κανόνων. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα έχει το λόγο η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ. πολύ, κύριε. Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε αυτό το κοινό ψήφισμα. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αφαιρεί από τις χώρες μέλη το δικαίωμα και τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται μεταξύ τους ως ισότιμοι εταίροι για σημαντικά οικονομικά θέματα. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κρίση θα πρέπει να κερδίσουμε εκ νέου την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η αναζήτηση νέων τρόπων ε, ε, δανεισμού ε, όλα αυτά μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μοδόδρομος προς μια νέα υπερχρέωση, μια δόση προς την κόλαση και αυτό ισχύει και για την επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ζαμπόρσκα και τώρα συνεχίζουμε με την έκθεση του κυρίου Φλόρεντς. Ο κύριος Χάνν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με εξέπληξε το ύφος των παρατηρήσεων που έχουν εκφραστεί εδώ, σε αυτή την αίθουσα, από τότε που έλαβε χώρα η τελευταία σύνοδος, αναφορικά με τη Βρετανική στάση. Ε, περιφρονητικό τρόπο μας σχολιάζουν. Εγώ θεωρώ όμως ότι είναι μια επικοδομητική βάση διαπραγμάτευσης. Αφού δεν θα συμμετάσχουμε εμείς σε αυτή τη νέα συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι λογικό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι το φόρουμ για περισσότερη εναρμόνιση π.χ. φορολογίας, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης για μεγαλύτερη ε, πολιτική ενοποίηση. Βέβαια, αν αφαιρέσουμε περιεχόμενο και κρατήσουμε το φλοιό, θα έχουμε ένα ε, τσόφλι κενό. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι. Μπορεί να, ε, μπορεί να χάσετε λοιπόν έναν ε, ενοχλητικό κάτοικο της πολυκατοικίας, αλλά μπορεί να κερδίσετε έναν ευπροσίγουρο γείτονα στη διπλανή πολυκατοικία. Ο επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια είδαμε να Αυξάνεται ο οικιακός εξοπλισμός των πολιτών. Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία για να ικανοποιήσει τη ζήτηση για προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας. Ο ηλεκτρικός οικιακός εξοπλισμός έχει μικρό κύκλο ζωής, απαξιώνεται γρήγορα και επομένως πρέπει να εξετάσουμε την απόρριψη αυτού. Θα πρέπει να ανακυκλώνεται σωστά. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τη στρατηγική της Επιτροπής για το 2020. Καλό τους διανομής και προμηθευτές λιανικής να έχουν όλο και περισσότερα ε, σημεία υποδοχής όλων αυτών των ε, οικιακών ηλεκτρικών μηχανημάτων. Το περιβάλλον ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα και οφείλουμε στους πολίτες μας να τους εξασφαλίσουμε ένα καθαρό περιβάλλον σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Τάνο και κυρία Πιετικάνεν. Συμφωνώ απολύτως με αυτήν την νομοθεσία που θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιτύχουμε τους στόχους που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη ε, θέλει να επιτύχει στα πλαίσια της στρατηγικής ε, για τις πρώτες ύλες λείπουν ε, πρώτες ύλες, λείπουν ε, κάποια μέταλλα, λείπουν πόροι λοιπόν ε, συνολικά και πιστεύω ότι αυτή η συλλογή <clears throat> των ηλεκτρονικών απορρίτων θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έλενα Μπασέσκου έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή γιατί θεωρώ ότι η τροποποίηση της οδηγίας θα επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές. Αναφέρομαι κυρίως στη μεθοδολογία της συγκέντρωσης και τις κατηγορίες ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Ένα άλλο σημαντικό θετικό στοιχείο είναι η έλλειψη στρατηγικών ε, πρώτων υλών, καθώς επίσης και η ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση στοιχείων. Η συμμετοχή των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων. Ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα. Ε, ας πούμε, στη χώρα μου υπάρχει μια, ε, ένα site ε, που δίνει πληροφορίες όσον αφορά την ανακύκλωση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών. Ε, και, το, και εδώ και δύο χρόνια ξεκίνησε μια ετήσια για μεγάλη συλλογή τέτοιων ε, συσκευών στην Ρουμανία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μεζάρος. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά είναι τα απόβλητα που πολλαπλασιάζονται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να μεριμνήσουμε για την ανακύκλωση, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά για να μην βλάψουμε και τη δική μας υγεία, την υγεία όλων των πολιτών. Είναι γνωστό ότι ανακτάται η πλειονότητα των υλικών που απαρτίζουν ε, τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό οικιακό εξοπλισμό. Μπορεί να συγκεντρώνονται βέβαια, αλλά δεν ανακυκλώνονται στο σύνολό τους. Πρέπει λοιπόν να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τον κόσμο. Η τωρινή οδηγία δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να επιμερίσουμε τις ευθύνες ως προς τη συλλογή, τη συγκέντρωση και την κατανομή επίσης των αποβλήτων. Θα πρέπει να γίνεται διαλογή στην πηγή, επιλεκτική συγκέντρωση και να ληφθεί υπόψη η τιμή του προϊόντος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μεσάρος, λέει ο Πρόεδρος. Ο, η κυρία Σβίσμπουργκ έχει το λόγο. Κοιτάξτε, αυτή η έκθεση για τα απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πετυχαίνει το σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ αυτού που πρέπει να αποφασίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτού που πρέπει να αποφασίζεται σε εθνικό επίπεδο. Ε, διατηρείται η τρέχουσα μεθοδολογία και έτσι μέχρι τα τέλη του 2013 μετά θα έχουμε έναν ενδιάμεσο στόχο και θα έχουμε και το φιλόδοξο στόχο του 65% από το 2020 και μετά τα κράτη-μέλη που φιλοδοξούν να φτάσουν στο στόχο του 85% μπορούν να το πράξουν. Καλωσορίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικουρήσει τι χώρες που παλεύουν να εκπληρώσουν τους στόχους αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό να αυξήσουμε το ποσοστό του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος ανακυκλώνεται. Αλλά δεν θα πρέπει η προσέγγιση να λειτουργεί κατηγορηματικά, μη δίνοντας ευελιξία στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να επιλέξουν τους πιο εφικτούς στόχους, ώστε να δείξουν πόσο δεσμεύονται έναντι της πραγματικότητας αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σβίνμουρ. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο τώρα. Ε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ το συνάδελφο κύριο Φλόρεντς για τη θαυμάσια δουλειά που έκανε σε αυτή την έκθεση. Έχω την αίσθηση ότι πραγματικά έκανε μια πολύ καλή δουλειά και αναγνωρίζεται από όλους τους ομιλητές αυτό το σάμα. Βεβαίω πρόκειται για ένα τεράστιο τομέα για μα, γιατί έχουμε όλο και περισσότερο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έρχεται στην αγορά και είναι σημαντικό να συλλέγεται σωστά και ε, να ανακυκλώνεται. Ε, υπάρχουν θέρμητες πρακτικές όπως η εξαγωγή προ τρίτε χώρες. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε μέσω τη πρόταση να βελτιώσουμε το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών ε, νομίζω ότι είναι, δεν μπορεί αυτό παρά να αποφέρει κέρδος για όλους τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τάνοκ για την έκθεση της Κρίστας Κλάς. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση κλάς όσον αφορά τη χρήση βιοκτώνων και τη διάθεση στην αγορά. Νομίζω ότι η πρόταση είναι εξισορροπημένη και νομίζω ότι διατηρούνται πολύ βασικοί ε, στόχοι. Η, διαδικασία για την επεξεργασία χημικών ε, δραστικών ουσιών και προβληματικών ουσιών ε, συνεχίζει να ισχύει. Νομίζω ότι θα πρέπει, είναι ουσιαστικό να αλλάξει. Νομίζω ότι οι απαιτήσει που έχουν ε, εισαχθεί ε, θα πρέπει να αυξηθούν, θα πρέπει να υπάρξει μια απλούστευση, θα είναι ένα θετικό βήμα. Η θέση ενό υποχρεωτικού μηχανισμού είναι επίση σημαντική, έτσι όπω την προτείνει η έκθεση. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν οι επικαλύψει μέσω ε, στι μελέτε, μελέτες, στις μελέτε και τι γενομικέ μελέτε. Νομίζω ότι με το, η έκθεση αυτή καθιστά πιο εύληπτο τον κανονισμό. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ελένα Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, υπερψήφισα την έκθεση αυτή γιατί τα προϊόντα τα με στοιχεία βιοκτώνα χρησιμοποιούνται και στην κλωστοϊφαντουργία και στα καλλιντικά και σε πολλές άλλες βιομηχανίες και επομένως η χρήση τους θα πρέπει να διαφθετηθεί σωστά. Ε, ε, χρειαζόμαστε απλουστευμένες διαδικασίες αλλά ταυτοχρόνως ε, υψηλό επίπεδο προστασίας όσον αφορά την υγεία. Διαπιστώνω ότι το κεντρικό σύστημα αδειοδότησης θα υπάρχει θετική επίπτωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, <clears throat> τα ε, η επισήμανση η οποία θα είναι αναλυτική όσον αφορά την χρήση βιοκτώνων θα προστατεύσει καλύτερα τους ε, καταναλωτές. Ε, συμφωνώ με την ε, προσοχή η οποία έχει δοθεί όσον αφορά την σορευτική, το σορευτικό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα δεν έχουν ληφθεί μέτρα. Πάντως είναι ένα βήμα προς τα εμπρός οι προτάσεις της Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Μπασέσκου. Ο κύριος Πίτερ Γιάρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι χώρες μέλη ε, σήμερα συμφώνησαν για μια αναδιάταξη του κανονισμού για τα βιοκτώνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει μια ευρωπαϊκή, θα υπάρξει μια ευρωπαϊκή αδειοδότηση, διαδικασία αδειοδότησης ε, και που θα πρέπει και οι μη Ευρωπαίοι ε, παραγωγοί να τηρήσουν τα υψηλά ευρωπαϊκά στάνταρτς αν θέλουν να πωλήσουν τα προϊόντα στην Ευρώπη. Από την άποψη της Γεωργίας είναι σημαντικό βεβαίως να είναι διαθέσιμα τα βιοκτώνα που να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι γεωργοί μα. Πιστεύω ότι επετέφθη ένα καλό συμβιβασμό για μια βιώσιμη χρήση των βιοκτώνων από τη μία και αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων από την άλλη ή περιορισμό των ενδεχόμενων κινδύνων. Βεβαίω, ε, το θέμα αυτό βρίσκεται υπό εξέλιξη και δεν είναι η τελευταία φορά που θα ασχοληθούμε με αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιάρ και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σουίνμπουρν. Η διατήρηση της χρήσης των υφιστάμενων προϊόντων και η απουσία εναλλακτικών δεν είναι σωστή. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία του ανθρώπου αλλά και του ζωικού βασιλείου. Πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διατηρηθεί στα πρότυπα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ε, να διατηρηθούν όλα αυτά τα όρια. Και χαίρομαι γιατί θα επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα προϊόντα αυτά και οι ανανεώσεις δεν θα μπορούν να ξεπερνάνε τα 10 χρόνια. Να επιτρέπεται η χρήση τους σε, με ελεγχόμενο τρόπο. Αυτό είναι το πιο σωστό Άλλωστε τα χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ουαλία, στην ε, περιφέρειά μου. Η ρυθμισμένη χρήση είναι προτιμότερη από την απαγόρευση, την πλήρη απαγόρευση. Και βεβαίως θα πρέπει οι οι κανόνες να ισχύουν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σβίνπερν. Προχωρούμε τώρα στην έκθεση Μποβέ να δώσω το λόγο στον κύριο Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Είναι μια βιομηχανία, ένας κλάδος της οικονομίας, ενεργειακά ενεργοβόρος θα έλεγα και αναγνωρίζονται πολλά από τα χαρακτηριστικά τους σε αυτή την έκθεση. Η νομοθεσία που εφαρμόζεται και ισχύει από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά κάνει τα αγροκτήματά μας λιγότερα ανταγωνιστικά. Και η έκθεση προσπαθεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό. Τα μέτρα που αποτελούν μέρος του σχεδίου νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το 2013 θα δυσκολέψουν πολλούς από τους αγρότες μας και θα ε, επιβαρύνουν χωρίς να χρειάζεται όλη αυτή τη βιομηχανία, όλο αυτό το κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα έπρεπε να μεριμνούμε να λαμβάνουμε μέτρα που θα έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα στο κλάδο. Ευχαριστώ. Κύριε Τάνοκ, το λόγο έχει η κυρία Πιέτη Κάινεν. Κύριε Πρόεδρε, όπως και για το θέμα των ηλεκτρικών ηλεκτρονικών αποβλήτων και εδώ τίθεται το ζήτημα των πόρων. Και αυτό για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ απολύτως με την πολύ καλή αυτή η έκθεση που δείχνει ότι χρειαζόμαστε μέτρα, χρειαζόμαστε δράση σε όλες τις φάσεις της διατροφικής αλυσίδας. Ε, ποιο σύστημα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και μια σειρά, ε, ένα σύνολο μέτρων εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρούμε ένα αποτελεσματικό σύστημα έτσι ώστε <clears throat> θα πρέπει όσο γίνεται πιο υγιεινά τρόφιμα να υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και βεβαίως συμφωνούμε ε, και με τους στόχους που τίθενται και φυσικά θα πρέπει να δούμε ε, και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου Μποβέ γιατί θεωρώ ότι στις γεωργικές αγορές ο μηχανισμός τιμών ε, θα πρέπει να ε, προβλέπει η ισότιμη και δίκαιη ε, κατανομή των εισοδημάτων. Εδώ υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης ε, και επιπλέον πρόβλημα είναι ε, η μείωση της αγοραστικής ικανότητας ε, των πολιτών με ταυτόχρονη αύξηση της συγκέντρωσης σε πολύ μεγάλες αλυσίδες. Οι γεωργοί, ειδικά σε ορεινές περιοχές, δυσκολεύονται περισσότερο και πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην μεταφορά των αγαθών και τη συντήρησή τους, χρεώνονται περισσότερο. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια αποζημίωση για τους γεωργούς αυτούς επίσης. Θα πρέπει να υπάρξει και αποζημίωση για τις, από τα διευθυντικά ταμεία για τις περιοχές αυτές. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με τη σημερινή έκθεση πρωτοβουλία τη Επιτροπή Γεωργία επισημαίνουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα ε, πρόβλημα στη Γεωργία. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το κόστο πολύ περισσότερο από τι ε, τιμέ ε, στη Γεωργία. Θέλουμε όμω θεμητέ προποθέσει για όλου του παραγωγού. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να παρέμβει η πολιτική όταν δεν ε, διαφυλάσσονται αυτές οι θεμητές προϋποθέσεις παραγωγής. Έχουμε πολλές αγροτικές μονάδες, έχουμε πολλές μεσαίες επιχειρήσεις και έχουμε ένα εξαιρετικά συγκεντρωτικό εμπόριο από την άλλη. Ε, άρα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες ενώσεις ε, εκπροσώπησης ε, συμφερόντων που να γνωρίζουν την κατάσταση στην αγορά. Και νομίζω ότι το υφιστάμενο δίκαιο για κατάχρηση δευτεροσπόσεις θέσης στην αγορά και το δίκαιο για τα καρτέλ θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κέλλη. Uh, ε, ναι, θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή. Η συζήτηση η οποία έγινε σχετικά ήταν εξαιρετικά καλή και στο τέλος της ε, μέρας αυτής ασχολούμαι με αυτό το ιδιαίτερο σημαντικό πρόβλημα γιατί το ζήτημα του κέρδους ε, των, ε, που επιτυχάνουν οι πολυεθνικές εταιρείες είναι πολύ σημαντικό ενώ οι παραγωγοί κερδίζουν ελάχιστα από την άλλη οι μικροκαλλιεργητές. Γι' αυτό θα πρέπει να θέσουμε ένα τέλος σε αυτές τις αθέμητες ε, πρακτικές ιδιαιτέρως όσον αφορά ορισμένους από αυτούς τομείς κλειδί. Γιατί θα πρέπει να παρέμβουμε διευθυντικά σε αυτή την κατάσταση ούτως ώστε να έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση όλων των καλλιεργητών μας. Και πραγματικά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί σήμερα είναι οι, οι μεγαλύτεροι όμιλοι αυτοί που ελέγχουν τα πράγματα και η κατάσταση αυτή δεν είναι ε, σωστή, ούτε δίκαιη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέλλη και τώρα θα περάσουμε στην έκθεση όσον αφορά τις ανισορροπίες στην αλυσίδα εφοδιασμού και θα δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Κέλλη. Ναι, ε, το θέμα αυτό είναι παρόμοιο με το προηγούμενο θέμα και πραγματικά θα ήθελα να πω και πάλι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα στο επίπεδο των παραγωγών και ιδιαίτερα να καταπολεμήσουμε τις πολυεθνικές εταιρείες ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ισότιμες συνθήκες για όλους τους ενεχόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέλλη. Τώρα έχουμε τη διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Χάναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το διάστημα ανέκαθεν ε, διήγηρε τη φαντασία πολλών που ονειρεύονται την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Θεωρείται ότι αν κατακτήσουμε ευρωπαϊκά το διάστημα θα επιβεβαιώσουμε τη θέση μας σε αυτό τον κόσμο. Άλλωστε με το σύστημα Γαλιλαίο ο πρόεδρος Σιράκ ήθελε υποτίθεται να ε, νικήσει τον υπεριαλισμό των ε, Αμερικανών και ήταν όνειρο πάντοτε ένας Γάλλος να πάει στο φεγγάρι και να, προσελινωθεί Το θέμα είναι που κατά πόσο θα μπορούσαν να τον φέρουν πίσω βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, στις τελευταίες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε, φάνηκε ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκοπεί από την κοινή γνώμη, μας περιφρονεί όλους εμάς τους πολίτες και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, παρόλο που επιμένει να ετενίζει τον έναστρο ουρανό ως να μην συμβαίνει τίποτα. Ευχαριστώ, ο κύριος που έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου δυστυχώς ο μιλητής. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή διότι όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκομίσει πολλά ωφέλη από αυτό το εγχείρημα. Θα βελτιωθεί η τεχνολογία του διαστήματος, κάτι το οποίο θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Έχουμε τους δορυφόρους GPS, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενισχυθούν για να βοηθήσουν όλους τους εποχούμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να διασφαλιστεί ότι θα δίδεται προτεραιότητα ε, στα πλοία που τη χρειάζονται γιατί βρίσκονται σε επίγουσες συνθήκες. Ε, να βελτιωθεί η μεταφορά των προϊόντων κατά επέκταση ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ενισχυθούν άλλωστε ε, πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες. Καλή η έκθεση το πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο να χρηματοδοτεί το GMES, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να βρει έξωθεν χρηματοδότηση και έτσι αυτό αποτελεί επιπρόσθετο βάρος σε περίοδους οικονομικής λιτότητας και είναι το μόνο αρνητικό στοιχείο της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ η κυρία Σβίνμπερν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση για τη διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταθέτει εύλογες προτάσεις σε ένα τομέα όπου μπορούν πράγματι να αξιοποιηθούν οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συγκεντρωθούν οι πόροι, θα ε, ε, συγκεντρωθεί όλο αυτό το ευφυές κεφάλαιο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσουμε και να προοδεύσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικός. Και από τη στιγμή που η έρευνα στο διάστημα τελικά βρίσκει καθημερινές εφαρμογές εφαρμογές. Ε, η ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία σε βάθος χρόνου και θα μας ε, και θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το σύστημα Γαλιλαίος αλλά και, στο το σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού στην Ευρώπη, το GPS. Είναι ένας τομέας όπου πραγματικά μπορούμε να δημιουργήσουμε και να απολαύσουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ. Η πρόταση Καρόνα για την αποφυγή σπατάλης τροφίμων. Ο κύριος Άνναν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δικτατορία του Λουκασέγκο στη Λευκορωσία περιγράφεται ως το τελευταίο απομεινάρι του σοβιωτικού καθεστώτος στην Ευρώπη. Όσοι το λένε αυτό όμως δεν έχουν υπόψη τους την ε, κοινοτική γεωργική πολιτική η οποία τόσο πολύ περιχαρακώνει την ελευθερία δράσης και τόσο πολύ πλήττει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην Αφρική από τη στιγμή ε, που πλήττει τόσο τους φτωχούς και δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία μας αντεβάζοντας τις τιμές, από τη στιγμή που προκαλεί στρέβλωση πρωτοβουλειών στην Ήπεθρο, από τη στιγμή που ε, πλήττει χώρες όπως η δική μου οι οποίες είναι καθαροί εισαγωγή τροφίμων. Ωστόσο, οφείλουμε να μελετήσουμε περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται μια συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι απαραίτητα αγρότες, γιατί οι πληρωμές έχουν αποσυνδεθεί από τη γη σε διάφορους φορούς δίνονται, σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή και άτομα ολόκληρα λαμβάνουν επιταγές τις οποίες εξαργυρώνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξαγοράσει την εμπιστοσύνη μια συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο καλύτερο μηχανισμό στην Ευρώπη για να γίνει αναδιανομή του πλούτου από του φτωχού στου πλουσίου. Και όλα αυτά τα λουζόμαστε τώρα με την ε, κρίση και τα οικονομικά προβλήματα. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, Υπερψήφισα τι αλλαγέ που θεσπίζει η έκθεση Καρόνα στην παρούσα κρίση και με έναν παγκόσμιο πληθυσμό να αυξάνει με τον παρόντα ρυθμό. Η σπατάλη τροφίμων θα πρέπει να μειωθεί γιατί ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερα. Οι βέλτιστε πρακτικέ και ένα καλύτερο συνδυασμό μεταξύ των χωρών μολών θα ήταν μια ενδεδειγμένη λύση. Νομίζω ότι ένα σημαντικό θέμα που επισημαίνει η έκθεση είναι ότι κανένα ε, που αφορούν ε, την πώληση κάτω από την ε, τιμή δεν έχουν ακόμα θεσπιστεί. Είναι σημαντικό οι ελληνικοί έμποροι να μπορούν να πολλούν τρόφιμα που είναι κοντά σε λήξη σε χαμηλές τιμές. Είναι σημαντικό σε χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένε χώρες υπάρχει απαγόρευση να πωλήσουν σε χαμηλότερε τιμέ οι λιανέμποροι. Νομίζω θα πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο συντονισμό μεταξύ των χωρών μελών για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και τέλο, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Χάνεν, ο οποίο ε, ζητάει μια πιο δραστική μεταρρύθμιση τη γεωργική πολιτική, κάτι το οποίο είναι καθοριστικό για το μέλλον. Ο κύριος Πίπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση με μεγάλη ευχαρίστηση γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 90 εκατομμύρια τόνοι ε, τροφών που μπορούν ε, να αναλωθούν καταλήγουν ε, στα σκουπίδια. Είναι πραγματικά αφόρητο το ίμιση των τροφίμων τελικά να καταλήγουν στα σκουπίδια. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. πρέπει να γίνει εκ της Κομισιόν μια ανάλυση για τα αίτια αυτής της κατάστασης. Και όταν εμείς ως καταναλωτές έχουμε την βασική ευθύνη για αυτή τη σπατάλη, θα πρέπει πραγματικά να αναπτύξουμε μια πολιτική σκέψη. Ένα βασικό θέμα είναι η διάρκεια λήξης των προϊόντων που τελικά οδηγεί σε υπερβολικά μέτρα και σε σπατάλη τροφίμων στην Πολωνία αντί για την ελάχιστη λήξη λέει ότι προτιμάται η ανάλωση μέχρι την τάδε ημερομηνία. Ε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε από τις χώρες εκείνες που πραγματικά αντιμετωπίζουν με ένα βιώσιμο τρόπο την ε, κατανάλωση τροφίμων. Η κυρία το Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου Καρόνα λαμβάνοντας υπόψη και τις προειδοποιήσεις ε, της ε, ΦΑΟ για τις ε, σημαντικές ανισότητες της παραγωγής τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε σωστή γεωργία που θα συνοδεύεται παράλληλα και από υπεύθυνη κατανάλωση. Αυτή είναι και η βάση της επιστημιστικής ασφάλειας. Θέλουμε ένα νέο θεμελιώδες δίκαιο και για τους πολίτες της Ευρώπης και για τους πολίτες του κόσμου. 180 κιλά ε, ε, ε, τροφίμων που καταλήγουν στο σκουπιδοντινή μετράει κάθε ένας Ευρωπαίος πολίτης ενώ υπάρχουν οικογένειες οι οποίες τρέφονται πάρα πολύ άσχημα και υπάρχουν ορισμένες περιοχές της Ευρώπης όπου η κακή διατροφή των παιδιών είναι από τις υψηλότερες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πίτερ Γιάρ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη βδομάδα ασχολήθηκε με ένα πολύ σημαντικό θέμα, δηλαδή τη σπατάλη των τροφίμων. Και πραγματικά αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερω, γιατί στι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό αφορά το ίμιση τη των τροφίμων. Δηλαδή τα τρόφιμα δεν καταλήγουν εκεί όπου ανήκουν ε, στον καταναλωτή για να αναλωθούν, αλλά πετιούνται στα σκουπίδια και θα ήθελα να συμπληρώσω τον κύριο Πίπερ ότι, που είπε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι παραπάνω, έχουμε κάπως καλύτερες ιδέες. Ε, έχει δίκιο. Ε, η έκθεση είναι καλή, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά αποδεκτές και αποτελεσματικές δράσεις. Και θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο με ε, εξοργίζει αφορά την ημερομηνία ε, λήξης των ε, προϊόντων ε, το θέμα αυτό. Θα πρέπει εδώ η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα, μάλλον τα τρόφιμα τα οποία δεν μπορούν να αναλωθούν από τον άνθρωπο, τουλάχιστον να χρησιμοποιούνται τα τρόφιμα αυτά για ζωοτροφές. Αυτή είναι η πρόταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, της πίεσης που ασκείται στους καλλιεργητές να χρησιμοποιήσουν περισσότερα ε, ε, τρόφιμα με λιγότερα χρήματα, η έκθεση μοιάζει σωστή. Ωστόσο, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει στα 9 τρισεκατομμύρια το 2050. Είναι λογικό λοιπόν να μειώσουμε τη σπατάλη των ε, τροφίμων ως μέρος στρατηγικής εφοδιασμού με τρόφιμα. Ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα δίκτυο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνη και βέλτιση των πρακτικών όσον αφορά τη μείωση τη πατάλη. Θα πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα την έρευνα και να βελτιώσουμε τι τεχνολογίε για την επεξεργασία των ε, βιολογικών αποβλήτων υπάρχει η ανάγκη βιομηχανία να διαδραματίσει εδώ ένα καθοριστικό ρόλο και να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συσκευασία που θα πρέπει να γίνουν καινοτόμε ε, προτάσεις. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ανταγωνιστική αγορά η οποία να διαθέτει τα τρόφιμα με έναν οικολογικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αλλά δεν θα πρέπει να αντικαθιστούμε τις λύσεις που δίνει η ίδια η αγορά με έναν υπερβολικό φόρτο ενωσιακών κανονισμών. Ο κύριος Κούκαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της πατάλης των τροφίμων είναι ένα όλο και αυξανόμενο ευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο αντανακλάται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού με τρόφιμα. Και θα ήθελα λοιπόν να χαιρετήσω την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση της σπατάλης το 2020. Ελπίζω ότι η έκθεση που εγκρίναμε σήμερα και εγώ την υπερψήφισα θα συμβάλλει προς την εκπλήρωση αυτού του στόχου. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο Επίτροπος κ. Ποτότσνικ ότι πρόσφατα όπου πολλές χώρες πάσχουν από έλλειψη τροφίμων, στην παρούσα κατάσταση σε πολλές ε, χώρες πάσχουν από έλλειψη τροφίμων, η σπατάλη τροφίμων στην Ευρώπη είναι ηθικά απαράδεκτη. Ε, νομίζω ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα όχι μόνο για τις αίτιες, και τα αποτελέσματα της σπατάλης αλλά και για τους τρόπους μείωσης αυτής της σπατάλης. Θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω το αίτημα του Κοινοβουλίου να ανακηρύξει το έτος 2013 έτος καταπολέμησης της σπατάλης σαν ένα εργαλείο συνειδητοποίησης του πληθυσμού προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κούκαν. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν έκανα την έρευνά μου για το ζήτημα αυτό, πρέπει να σας πω ότι με εξέπληξαν οι αριθμοί ο αριθμός των οικοκυριών που σπαταλά τρόφιμα αξίας χιλίων ευρώ ετησίως είναι τεράστιος και το ποσό αυτό είναι πολύ μεγάλο. Κάτι πρέπει να γίνει. Τα στατιστικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Το 60% των τροφίμων που πετάγεται είναι βρόσιμο και το βασικό, βασικός λόγος γι' αυτό είναι η σύγχυση σε σχέση με την ετοκετοθεσία, με τη, με τη Θα πρέπει να ενημερώσουμε καλύτερα τον κόσμο και να λάβουμε υπόψη μας και τις εκπομπές που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή των τροφίμων και να κοιτάξουμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ε, σωστή ε, βιολογική διαχείριση των τροφίμων που ε, πετιόνται. Πολλή δουλειά έχουμε να κάνουμε λοιπόν. Ευχαριστώ τελευταίος ο κύριος Ρέπο παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου μιλητής δυστυχώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ διότι εκλεγήκατε εσείς ε, προσωπικά πρώτος αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση για την καταπολέμηση της πατάλης των τροφίμων. Πάρα πολλοί Ευρωπαίοι διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, αγωνίζονται να επιβιώσουν, ενώ από την άλλη πάρα πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο ε, πάσχουν από υποσυτισμό. Αυτά είναι δεδομένα. Και εμείς στην Ευρώπη πετούμε 120 κιλά ε, τροφίμων ε, ανά άτομο. Τρόφιμα τα οποία είναι απολύτως βρόσιμα κάτι το οποίο έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στο, σε περιβαλλοντικό επίπεδο, αλλά και κάτι το οποίο από ηθική σκοπιά είναι πολύ ε, επικριτέο, θα έλεγα. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα αυτό. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για τρόφιμα τα οποία είναι απολύτως βρόσιμα. Είναι απολύτως ανόητο σε οικονομικό επίπεδο. Είναι σαν να πετούσαμε χάρτονομίσματα στον σκουπιδοντενεκέ. Ευχαριστώ κύριε Ρέπο. Έχω πάρει από το Συμβούλιο τις θέσεις που έχουν εγκριθεί από τη, στην πρώτη ανάγνωση ε, και ε, έχουν γίνει δεκτά, ε, επομένως οι τίτλοι θα